υπάρξει ένας διάλογος για ένα τόσο σημαντικό θέμα και να συνεχιστεί με τους νέους συνομιλητές μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Ολοκληρώνοντα αυτή τη συζήτηση, πέντε προτάσει ψηφίσματο κατατέθηκαν από πέντε διαφορετικέ κοινοβουλευτικέ ομάδε. Του πράσινου, της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών, το, της Συμμαχίας των Φιλελευθέρων, της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Λαϊκού Κόμματος και Συνομοσπονδιακής Ενωτικής Αριστεράς. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε έτσι. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Αξιότιμοι συνάδελφοι, η επόμενη συνεδρίασή μας θα διεξαχθεί αύριο, 5η, 7η Απριλίου, από τις 9 στις 1 και μετά από τις 15 έως 17.00 έχει δημοσιευθεί η μερίσια διάταξη και είναι και στην ιστοσελίδα του Ευρωκοινοβουλίου διαθέσιμη. Λίγη συνεδρίαση. Εύχομαι σε όλους καλή νύχτα. Γεια σας.